και εσείς όπως και εγώ. Ας περάσουμε αμέσως στις ψηφοφορίες. Έκθεση της κυρίας Γκέριγκερ. Η ημερήσια διάταξη λοιπόν, σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία, έκθεση της κυρίας Γκέριγκερ, τίθεται σε ψηφοφορία, ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι. πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. Συγχαρητήρια στην κυρία Γκέριγκερ. Περνάω στην έκθεση Μπινεφ, πάντα με την συγκεκριμένη απλοποιημένη διαδικασία. Θέτω σε ψηφοφορία την έκθεση ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Συγχαρητήρια κύριε Μπινεφ. Τώρα περνάμε στην έκθεση Winkler. Πάντα με την απλοποιημένη διαδικασία ξεκινάει η ψηφοφορία ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι. πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή με μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια στον κύριο Βίνκλα. Έκθεση τώρα Χούμπνερ. Τίθεται σε ψηφοφορία ονομαστική κλίση. Τέλος. Και εδώ μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια. Κάποιος έχει στήσει το λόγο. Δυστυχώς ο μηχανισμός ψηφοφορίας μου δεν λειτουργεί. Θα το λάβουμε υπόψη, λέει ο Πρόεδρος. Έκθεση Σούριαν. Πάντα με την απλοποιημένη διαδικασία. Τίθεται σε ψηφοφορία η έκθεση Σούριαν. Εδώ απαιτείται ειδική πλειοψηφία. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίες. Και εδώ υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια λοιπόν στον κύριο Σούριαν. Έκθεση Ράπκαη. Ζητάει το λόγο ο κύριος Ουσπάκητς. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, δέχομαι πολιτική επίθεση. Πρέπει να σας πω ότι είμαι θύμα, επισήμως αναγνωρισμένο, θύμα πολιτικής επίθεσης. Το τμήμα Ασφαλείας συγκεκριμένα που έχει ε, πολιτικοποιηθεί στην ε, Λιθουανία προσπάθησε να με απαγάγει συγκεκριμένα στη διάρκεια της νύχτας. Δεν κατάφερα να συναντήσω τους ψηφοφόρους μου, κατάφερα όμως να πάω στην Ταϊλάνδη, στην Ινδονησία. Και ο συντάκτης των εκθέσεων ε, σας, της έκθεσης σας καλεί να παίξετε κι εσείς το ίδιο παιχνίδι. Πρέπει να ολοκληρώσετε σας έδωσα εκτάκτος τελείως το λόγο. Παρακαλώ, η συζήτηση έχει γίνει, δεν θα ξαναγίνει στην Ολομέλεια, σας ζητώ να κλείσετε. Δεν ε, έχω ομιλήσει καθόλου. Αντιθέτως, στην Επιτροπή ούτε καν μου δόθηκε ο λόγος και δεν μπόρεσα να σχολιάσω την απόφαση αυτή. Ούτε στη σταλινική εποχή να ήμασταν. Ονομαστική. Α, μάλλον όχι ονομαστική κλίση. Ποιοι είναι υπέρ της έκθεση Ραφκάη. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτή η έκθεση Ραπκάη. Έκθεση τώρα για Κολίνο. Για τη συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία. Ο κ. Γιακολίνο έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαι ιδιαίτερο σύντομο. Είναι η πρώτη συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία έχει πλέον ε, συμβολική σημασία. Πρόκειται για σημαντικές δραστηριότητες οι οποίες θα ενισχύσουν την παρέμβασή μας κατά της οργανωμένης εγκληματικότητας Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τις διαφορετικές ανάγκες ε, οι οποίες ε, υπάρχουν στις χώρες μας και στην Ιαπωνία και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει δεκτή η έκθεση αυτή. Είναι όπως είπα ένα θετικό βήμα έτσι ώστε να εξυγχρονιστεί η λειτουργία της δικαιοσύνης και μέσα από τις διμερείς σχέσεις. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Τίθεται σε ψηφοφορία η έκθεσή σας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η έκθεση γίνεται δεκτή. Συγχαρητήρια κύριε Γιακολίνο. Έκθεση Λέχνερ. Θέτω σε ψηφοφορία την έκθεση Λέχνερ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έκθεση Σρέντερ. για την βελτίωση της απασχόλησης. Έχει το λόγο η συγγήτρια, κυρία Σέντερ. Σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή στην οποία φτάνει αυτή η ψηφοφορία. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λάβαμε την πρωτοβουλία για μια ε, πρωτοβουλία για τις πράσινες θέσεις απασχόλησης και θέλουμε ε, να δώσουμε ε, ένα καλύτερο μέλλον στις αηφόρους θέσεις απασχόλησης για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση που θα έχουν σχέση με το, ε, την οικολογική διαμόρφωση του μέλλοντος με το Blue Act στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Κοινοβούλιο εργάστηκε σκληρά για την γνωμοδότηση αυτή και θα ήθελα ε, όλους τους εισηγητές ε, και τους κοιόδης εισηγητές που συνεργάστηκαν να τους ευχαριστήσω θερμά και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι διότι η Βελγική Προεδρία ανέφερε ήδη εκ των προτέρων ότι αυτή η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα τύχει συνέχεια και είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία και για το Συμβούλιο, τόσο ώστε να μπορεί να συμπεριληφθεί κάτι και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, τη διάσκεψη κορυφή. Και αυτό είναι ε, μια πρωτοβουλία πάρα πολύ σημαντική από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Θέτω σε ψηφοφορία διαντάσσεω χειρό ποιο είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και σας συγχαίρουμε, κυρία Σρέντερ. Έκθεση τώρα Τρατσκόφσκι. σε ό,τι αφορά την Ελβετία συγκεκριμένα και τα εμπόδια προ την πλήρη υλοποίηση εσωτερική αγορά σε όχα Ελβετία. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, ζητώντα τον έσω όσο το δυνατόν πιο τηλεγραφικό. Δεν δουλεύει. Α, ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο τη Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, τον κύριο Μάλκομ Χάρμπορ, ο οποίος ηγήθηκε όλου του ζητήματος, αλλά και τους σκιώδη συζητητέ ε, που είχα υποδειγματική συνεργασία μαζί του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία δυνατάσεω τη χειρό. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απόχέ. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια έκθεση Ζάλμπα Μπιντεγκάινα για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Κορέας και τη ρήτρα, μερή ρήτρα διασφάλισης. Ψηφοφορία ομαδών των τροπολογιών. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Όλες οι τροπολογίες θέτω σε ψηφοφορία τώρα την τροπολογημένη πρόταση της Επιτροπής είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Σύμφωνα με τον κανονισμό τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την ε, Νότια Κορέα νομίζω θα διανοίξει πολλέ δυνατότητε και για την ευρωπαϊκή και για την κορεατική βιομηχανία. Για να μην υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα όμω για την ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία, θα πρέπει να υπάρχει μια αποτελεσματική ρήτρα διασφάλιση. Όλε οι πολιτικέ ομάδε ομόφωνα την προηγούμενη εβδομάδα αποφασίσαμε ότι έφτασε η ώρα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποφασίσει για τι ε, τροπολογίε που 27 ψήφοι πέρ τη και μόνο μία ψήφο κατά περιεξε στην αρμόδια επιτροπή τον Ιούνιο. Είναι πολύ σημαντικό ε, να υπάρχει η απαραίτητη αποτελεσματικότητα στη ρήτρα διασφάλισης. Ε, θα ψηφίσουμε μόνο τις τροπολογίες, όπως ξέρετε, και με βάση με τον κανόνα 57 προ προτείνουμε αναβολή τη πληροφορία για την έκθεση νομοθετικού περιεχομένου για τη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Αποφασίσαμε επίσης ομόφωνα να μην κλείσουμε την πόρτα σε μια ενδεχόμενη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση που θεωρούμε ότι είναι εφικτό να επιτευχθεί. Βέβαια, ε, θέλουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ενότητας, ε, δύναμης όλων των πολιτικών ομάδων και εξού και η σημασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά να στηρίξει με αποφασιστικότητα όλο το πακέτο τροπολογιών. Ευχαριστώ. Η πρότασή σας ήταν σαφής. Έχει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, Όπω είπε και ο Επίτροπο Δεχούχτ χθε, χαιρετίζουμε την ε, εποφελή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Εμεί ε, αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε μια ψηφοφορία που αφορά μόνο τι ε, τροπολογίε και όχι την έκθεση για την κατάληξη σε συμφωνία ίσως και σε ε, πρώτη ανάγνωση. Ε, είχαμε στα τέλη Αυγούστου την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και στα μέσα τώρα θα έχουμε τη δεύτερη ε, διαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε δημοσίω να εκφραστούμε γιατί θέλουμε ο τριμερής διάλογος να διαδραματίσει το ρόλο του. Θα τοποθετηθούμε και θα εκφραστούμε και θα αναλάβουμε δεσμεύσει ή δυνατόν, μάλλον αν καταστεί αυτό αναγκαίο, στην ώρα της ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Περνάμε στην ψηφοφορία της πρότασης του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Η πρόταση γίνεται δεκτή. Τώρα για την έκθεση Μποβέ. Για την σωστή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων για τους γεωργούς. Τροπολογία 1. διανατάσσεως των χειρών. Η ψηφοφορία ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ένα απορρίπτεται. Θέτω σε ψηφοφορία τώρα την παράγραφο 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 6 γίνεται δεκτή. Θέτω τώρα σε ψηφοφορία την 8 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. Στην παράγραφο 10. Πάντα σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Παράγραφος 13. Α. Θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 10. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίας. Αυτή τη φορά είχα δίκιο. Λοιπόν, στην παράγραφο 13. Ονομαστική κλίση. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίες. Η παράγραφος αυτή απερίφθη. Προτείνεται μια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 21. Κόστιγκερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην παράγραφο 21 χρειάζεται συμπλήρωση των λέξεων για τα γεωργικά προϊόντα να λέει το κείμενο το οποίο λέει τα εξή. Θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να απαγορεύεται η πώληση σε πολύ χαμηλέ τιμέ γεωργικών προϊόντων, σε τιμέ κάτω του κόσμου. Λοιπόν, είναι κάποιο κατά αυτή τη προφορική τροπολογία. Δεν νομίζω. Συνεπώς συνεχίζουμε. Παράγραφος 21. Ονομαστική κλίση. Ξεκινάμε. 21. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Η 21 γίνεται δεκτή. Παράγραφος 24. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά Αποχές δεκτό. Παράγραφος 25. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεκτή μάλλον. 28 παράγραφος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 33. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά Αποχές δεκτή. 34. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Παράγραφος 36 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα 36 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Παράγραφος 37 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, για μια στιγμή για μια στιγμή. Έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάμε για το πρώτο τμήμα της 37. Πέρας ψηφοφορίες. Δεκτό το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα. Ξεκινάμε. Τέλος ψηφοφορίας. Δεκτό το δεύτερο τμήμα. Το τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορία. Και το τρίτο τμήμα γίνεται δεκτό. Παράγραφος 38 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Το δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Παράγραφος 39 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. 41. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η 41. 42 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Α. Καλώς θα υπάρξει λοιπόν ηλεκτρονικός έλεγχος για την 41. Ξεχωριστή ψηφοφορία για τις 41. Πέρας ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτή. Τελικά γίνεται δεκτή. 42 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Παράγραφος 46 πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτό. 47 πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα του 47 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτό. 52. Ονομαστική κλίση για την 52. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 54 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Παράγραφος 60. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 61. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 62. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 64. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Καλός ηλεκτρονικός έλεγχος στην 64. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Στο L λατινικό ποιοι είναι ε, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Στο μήλα την οικοπή είναι υπέρ. Κατά. Δεκτό. Θέτω τώρα το σύνολο του ψηφίσματος. Σε ψηφοφορία ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συγχαρητήρια στον κύριο Μπούβε. Περνάμε τώρα στην έκθεση πόρτας για την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής. Θέτω σε ψηφοφορία την παράγραφο 16 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Τρίτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Η πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συγχαρητήρια στον κύριο Πόρτας. Περνάω τώρα στην έκθεση ΣΒΙΦΚΑ για τη διεθνή δικαιοδοσία και εκτέλεση αποφάσεων σε ε, υποθέσεις εμπορικές και αστικές. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέτω σε ψηφοφορία τώρα την πρόταση ψηφίσματος της Αρμόδιας Επιτροπής ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συγχαρητήρια στον κύριο Σβίφκα. Έκθεση Παρφάνοβα. Παράγραφος 2. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 8 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την παράγραφο 8 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίες. Απερίφθη η παράγραφος 8. Παράγραφος 9 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. Λοιπόν, παράγραφος 11. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Λοιπόν, ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 11 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτή. Παράγραφος 18. Σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 18. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτό. 21. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 23. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 12. Ποιοι είναι υπέρ. Δεκτό. Το Ι τα λατινικό ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Το Ι λατινικό ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Στο έλα ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Στο όμικρον σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Στο S λατινικό ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Στο σύνολό του το ψήφισμα τώρα. Α, συγγνώμη, δεύτερο τμήμα του S. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία Παρβάνοβα. Περνάμε τώρα στην έκθεση ποιετικά είναι για το ρόλο των γυναικών. Θέτω σε ψηφοφορία την παράγραφο 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Παράγραφος 10. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Παράγραφο 28. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά Δεκτό. Παράγραφος 33. Το σημείο 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Παράγραφος 35. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Το σύνολο της προτάσεως ψηφίσματος. Ονομαστική κλίση. ποιέτικα είναι. Ψηφίζουμε. Τέλος της Μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια. Κύριε Πιετικάινεν. Λόκεγκαρντ. Έκθεση Λόκεγκαρντ. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Ψηφίζουμε τώρα στο σύνολό της την έκθεση. Όχι. Δεν υπάρχει λόγος μου λένε οι Κλείσαμε τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Επεξηγήσεις ψήφου. Καλή όρεξη σε όλους.